κατατέθηκαν και έχουν υποβληθεί και 7 συμβαστικέ τροπολογίες από τον εισηγητή. Θα ήθελε ο εισηγητή το λόγο. Αν όχι, θα πρότεινα να περάσουμε ευθύ αμέσω στην ψηφοφορία. Να ρωτήσω όμως, πρωτού προχωρήσουμε, έχετε όλοι μαζί σας τις κάρτες σας. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που ίσως ξέχασε την κάρτα ψηφοφορίας του. Όχι από ό,τι φαίνεται. Είστε όλοι εξοπλισμένοι. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Επειδή έχουμε πολλούς νέους συναδέλφους, να πω ότι ψηφίζουμε επί των ε, τροπολογιών διανατάσσεως της χειρός και τις συμβαστικές τροπολογίες θα τις ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Και όποτε δεν υπάρχει σαφήνεια ως προς το ποιο είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διανατάσσεως της χειρός, τότε επίσης θα ελέγχουμε την ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι είναι σαφές, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με την τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές. Αυτό θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε, συνάδελφοι, επί της τροπολογίας 4 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. So. Jetzt ist die Abstimmung eröffnet. Ich schließe. Πέρας της Dieser Änderungsantrag ist abgelehnt. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία α. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Schließe die Abstimmung. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Η συμβαστική τροπολογία εγκρίνεται. 45 υπέρ, 0 κατά, 0 αποχές. Περνάμε στην τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι καλό θα είναι να το ελέγξουμε αυτό ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Επί της τροπολογίας 14, άρχιτη ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Α, όχι, ήταν αρκετά σαφές το αποτέλεσμα. 38-7. Ε, συμβαστική τροπολογία Β. Και πάλι ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. Schließe die Abstimmung. Πέρας της Εγκρίνεται. Με μεγάλη διαφορά. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία σε Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Schließe die Abstimmung. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Συμβαστική τροπολογία D. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Schließe die Abstimmung. Πέρας της ψηφοφορίας. zu schnell. klar angenommen. Wir fahren mit... Εγκρίνεται. 32. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ, Κατά. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να το ελέγξουμε αυτό ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Schließe die Abstimmung. Πέρας της ψηφοφορίας. Dieser Antrag ist abgelehnt. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ε. Άρχεται η ψηφοφορία. σλίσε Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται ομόφωνο. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται επίσης ομόφωνα. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να το ελέγξουμε αυτό ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ επί της τροπολογίας 48 τώρα Ich schließe die Πέρας της απορρίπτεται Τροπολογία 49. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 51. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, ζητήθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία για έλεγχο. Οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα επί της τροπολογίας 52. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία, την οποία επίσης παραδοσιακά κάνουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία επί του συνόλου της γνωμοδότησης. Πέρας της ψηφοφορίας. Α, το πήγα λίγο γρήγορα. Εντάξει, περιμένουμε λίγο ακόμα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίζετε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 39 υπέρ, 5 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Και... Πάμε τώρα στα επιμέρους έργα. Τροπολογία 6001. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 6002. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ε, τροπολογία 6000 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 60-20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 60-25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, καταπίπτουν οι επόμενες, συνεχίζουμε με την 6024 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 60-23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 60-42 υπέρ κατά αποχές. Αυτό θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Επί της 6042. Πέρας. Δεκτή 24 προς 21. Άρα Πάμε τώρα στην 6032. υπέρ. 60-32 ε, Κατά αποχές δεκτή. 6018. υπερ Κατά αποχές δεκτή. 60-30 υπέρ κατά αποχές αυτό χρειάζεται ηλεκτρονικό έλεγχο ψηφίζουμε την 60-30 ηλεκτρονικά πέρασε αυτή απερίφθη. 60-13 υπέρ κατά αποχές απορριπτεται σαράντα πέντε. υπέρ κατά αποχές δεκτή. 60-45 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Πάμε τώρα στην 60-34. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος δεν είχα μεγάλη συμμετοχή ψηφίζουμε την 6034 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας σαφώς δεκτή 6007 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60-35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60-19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6.038 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Άρα ψηφίζουμε την 6006 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 6017 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 6041 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 6014 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60-44 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 60 6004 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές εδώ χρειάζεται έλεγχος Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η τροπολογία γίνεται δεκτή. 60-27 υπέρ, κατά, αποχές και αυτή γίνεται δεκτή. 60-39 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Δεν έχουμε τελική ψηφοφορία φυσικά, αυτά είναι επιμέρους θέσεις του προϋπολογισμού. Εδώ συγχαίρουμε την τον εισηγητή. Θέλει να λάβει το λόγο ο εισηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και να σας υπενθυμίσω ότι στη γνωμοδότηση αποφύγαμε περικοπές στο γεωρικό προϋπολογισμό. Αυτό επιθυμούμε ως Επιτροπή Γεωργίας να διαφυλάξουμε αλόβητο το γεωρικό προϋπολογισμό. Και ελπίζω να ληφθεί υπόψη διόντως η γνωμοδότησή μας από την αρμόδια καθήλη Επιτροπή που είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Τώρα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα της δυνατότητας κατοχύρωσης των φυτών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με σκοπό την υποβολή γραπτής δήλωσης στο Διευρυμένο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Αυτή είναι η υπόθεση G3 19. Ε, ζητήθηκε ε, από τον συνάδελφο Χούιτεμα να γίνει Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που το θέσατε στην ημερήσια διάταξη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Πού έγκυται το πρόβλημα. Το 2015 δύο ποικιλίε φυτών ε, έλαβα δίπλωμα βριστέχνιας Ε, μία ποικιλία πιπεριάς και μία άλλη. Με κλασική βελτίωση ε, μέθοδο, μέθοδο βελτίωση φυτών. Μια βιολογική διαδικασία δηλαδή, που είναι φυσιολογική διαδικασία της βελτίωσης των φυτών. Γιατί είναι επικίνδυνο όμω το θέμα αυτό. Δεδομένου ότι μια ποικιλία φυτών, για παράδειγμα το κόκκινο χρώμα στις ντομάτες θα καλυφθεί, θα κατοχυρωθεί από δίπλωμα ευρυστεχνίας, θα ανήκει σε μια ε, συγκεκριμένη εταιρεία. Οπότε οι υπόλοιποι βελτιωτέ φυτών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το κόκκινο χρώμα. Οπότε αυτή η εταιρεία που έχει το δίπλωμα θα έχει και το μονοπόλιο λαχανικών και φρούτων. Κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο και θα αφήσει γενετικό υλικό φυτών στα χέρια μερικών μόνο εταιριών. Το 2015 λοιπόν μαζί με κάποιους συναδέλφους από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία ενός ψηφίσματος που υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία και απαγορεύει τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για ε, ποικιλή φυτών που είναι αποτέλεσμα μιας κλασικής βιολογικής διαδικασίας βελτίωσης. Και στο Συμβούλιο όλα τα κράτη-μέλη στήριξαν το ψήφισμα και εξέφρασαν την ανησυχία τους ε, ε, σε περίπτωση που δοθούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας για βιολογικές διαδικασίες στη βελτίωση των φυτών. Και μάλιστα και Επιτροπή δήλωσε ότι ήταν μια λαθασμένη ερμηνεία της σχετικής οδηγίας ε, ε, ε, που δεν επιθυμούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα κατοχήρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνία βιολογικών διαδικασιών βελτίωση των φυτών. Και μάλιστα το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα διευκρινιστικό σημείωμα δηλώνοντας ότι δεν επουδενή η πρόθεση των νομοθετών να χορηγηθούν τέτοια διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις εταιρείες. Και μάλιστα και το Συμβούλιο του, γραφείου, του Ευρωπαϊκού Γραφείου ήταν τη ίδια γνώμη ότι δεν θα πρέπει να χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνία σε τέτοια περίπτωση. Βέβαια, δεν είναι σαφές ε, στο σχετικό κείμενο. Στον εφαρμοστικό κανονισμό υπάρχει, αλλά όχι στη σχετική σύμβαση. Ε, βέβαια, το Τεχνικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία λέει ότι η σύμβαση δεν είναι αρκετά ξεκάθαρη και σαφής, ότι δηλαδή απαγορεύεται η κατοχήρωση με δίπλωμα ευρυστεχνίας ε, ποικιλιών φυτών που είναι αποτέλεσμα μιας βιολογικής διαδικασίας βελτίωσης. Γι' αυτό ε, όταν καλέσαμε τον ε, Πρόεδρο το συζητήσαμε και υπάρχει μια ιεραρχία της για την λήψη της απόφασης για τη δυνατότητα κατοχύρωση ή όχι. Το διευρυμένο Προεδρείο είναι υπεύθυνο. Και Εμεί ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητούμε και από την Επιτροπή Γεωργίας ε, να συντάξουμε ένα νέο ψήφισμα ώστε και ε, το νέο κοινοβούλιο και οι νέοι ευρωβουλευτές να στηρίξουμε την ψήφο του αυτή την άποψη. Ότι δηλαδή δεν είναι σωστό να χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας για ποικιλίε φυτών που είναι αποτέλεσμα μιας βιολογικής διαργασίας βελτίωσης. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Χόιτεμα. Η Κομισιόν τώρα έχει το λόγο. Στον κύριο Τζιπίνη από τη νομική υπηρεσία της Κομισιόν ε, που κάθεται, δεν βλέπω. Ονομάζομαι Χέρι Τσιπίνη από την νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα και σας ευχαριστώ που εγκύπτεται σε αυτό το σημαντικό θέμα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει δήλωση στο διευρυμένο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας με τη θέση που εξηγήσαμε και στη δήλωση του 2016, ότι δηλαδή προϊόντα που είναι ε, αποτέλεσμα βιολογικής διαδικασίας κυρίως και τέτοια φυτά δεν μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και οποιαδήποτε βοήθεια, συνδρομή, αρρωγή από την Επιτροπή σας με οποιαδήποτε μορφή είναι ευπρόσδεκτη. Και θα ήθελα να σας πω ότι το διευρυμένο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου έχει θέσει ως την 1η Οκτωβρίου καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τέτοιων δηλώσεων. Ελπίζουμε να στηρίξετε πλήρως το περιεχόμενο του σημειώματος του 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απαγορεύει τη δυνατότητα κατοχήρωσης σε τέτοιες περιπτώσεις από την DigiGrow, Grow, Mary Hoover. Εμείς είμαστε αρμόδιοι για το σημείωμα και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει αυτό το διάβημα προς το Διευρυμένο Συμβούλιο Προσφυγών του Γραφείου. Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις της Κομισιόν. Διάφοροι συνάδελφοι ζήτησαν ήδη το λόγο. Η κυρία Σράια Πύρικ, καταρχήν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Γιάνν Χαϊτεμα σας εξήγησε διεξοδικά την κατάσταση. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία είχαμε εκτενείς συζητήσει για το θέμα αυτό και ένα σχέδιο ψηφίσματος που μάλιστα εγκρίθηκε με πλειοψηφία. Δεν θα μακρηγορήσω, μακάρι να καταφέρουμε από κοινού να σημειώσουμε πρόοδο και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους αγρότες ότι είναι στο πλευρό τους. Γιατί φαίνεται ότι κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια δημιουργήθηκαν. Θα πρέπει τώρα να τα άρουμε επιτέλους. Ο κύριος Αντριέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Χαϊτεμα που επανέφερε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη με την ανταλλαγή απόψεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και το έχουμε ήδη συζητήσει. Αλλά είναι σημαντικό και οι νέοι να διευκρινίσουν τη θέση τους έχοντας γνώση του πράγματος. Εδώ μιλούμε για τη διπλώματα ευρεσιτεχνία σε βελτίωση φυτών που είναι αποτέλεσμα βιολογικής, φυσιολογικής βιολογικής διεργασίας. Μάλιστα, στυλιτεύσαμε την καταχρηστική χορήγηση διπλωματικών ευρεσιτεχνιών σε φυτικές ποικιλίε και το είπαμε αυτό και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Γραφείου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Είπαμε ότι μια τέτοια κατάσταση είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη και είναι μια καταχρηστική κατάσταση που ε, δίνει την ευκαιρία σε ισχυρέ εταιρείε ε, να λάβουν τέτοια διπλώματα ευρεσιτεχνία, ε, δημιουργώντας ένα μονοπόλιο de facto για φυτά. Είμαστε υπέρ της καινοτομίας και της κοινή χρήσης αυτής της καινοτομίας. Είναι λοιπόν μεγάλη ευθύνη πριν λήξει η προθεσμία των προσφυγών, η 1η Οκτωβρίου δηλαδή, να υποβάλουμε αυτή την γραπτή δήλωση. Δεν ξέρω αν επιληφθούν αργότερα και οι συντονιστές. Επήγε το θέμα και θα πρέπει ε, ρητά και κατηγορηματικά να επέμβουμε με τη δήλωση στο γραφείο στο, στο, στο Διευρυμένο Συμβούλιο Προσφυγών. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που ήδη είπαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Ρούιτεμα που, Κούιτεμα που έθεσε το θέμα ξανά και υποστηρίζω πλήρως την ιδέα του εδώ, δηλαδή να κάνουμε ψήφισμα ως Επιτροπή που απόλυτα ξεκάθαρα θα προβάλλει την απόψή μας. Γενικά αν δούμε όλο αυτό τον χώρο των βελτιωτών φυτών στην Ευρώπη, ε, θα δούμε ότι ε, θα, θα λέγαμε ότι είναι μεγάλη η παραγωγή. Όχι. Οι βελτιωτές, η παραγωγή νέων, δημιουργή νέων σπόρων είναι πάρα πολύ και μικρότεροι δημόσιοι στον τομέα της ε, γεωργίας δραστηριοποιούνται πολύ και για όλους αυτούς τους δημιουργούς σπόρων η ελεύθερη πρόσβαση στο γονιδιακό πουλ, αν θέλετε, στις τράπεζες που υπάρχουν, η ελεύθερη πρόσβαση εκεί, σε όλο αυτό το γονιδιακό υλικό, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν να κάνουν τις διασταυρώσεις και τις βελτιώσεις. Αν δεν γίνει αυτό, τότε η βελτίωση θα συνδυάζεται με υψηλότατο κόστος και έτσι θα εξοπεταχτούν από την αγορά οι μικροί δημιουργοί οι ε, μεγάλοι θα κατατροπώσουν τους μικρούς. Αυτό θα είναι ε, μια η δική μας κατάσταση στην Ευρώπη θα πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ, συνάδελφος Ταραμπέλα. Όντως, με κάλυψαν σε πολλά συνάδελφοι και ευχαριστώ τον κύριο Χαϊτεμέ για την πρωτοβουλία του. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήταν σαφέστατη ε, και με την διευκρινιστική της δήλωση του 2016 συμφώνησε με εμάς. Θα πρέπει να συσπηρωθούμε και να συγκεντρώσουμε μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ του νέου ψηφίσματος. Και μάλιστα στο Συμβούλιο Γεωργίας της 18 Μαρτίου το Βέλγιο ε, εξέφρασε την υποστήριξή του στο διευκρινιστικό σημείωμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2016. Και άλλε χώρε έκαναν το ίδιο. Οπότε και το Συμβούλιο είναι κατά πλειοψηφία υπέρ αυτής της θέσης, ώστε προϊόντα που είναι αποτελέσματα βιολογικών κυρίως διαδικασιών να μην δίνεται να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για να είναι διαθέσιμες όλες οι ποικιλίε σπόρων για όλους τους γεωργούς. Αυτό είναι δικό του συμφέρον και αυτή είναι η σημαντική μάχη που θα πρέπει να δώσουμε και είναι κρίμα που το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κάνει ε, από καιρού καιρών τέτοιε προτάσεις. Και αν όχι ομοφωνία, να επιδιώξουμε συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ του ψηφίσματός μας. Ευχαριστώ κύριο Χόισλινγκ. Ναι, είναι μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ, γιατί είχαμε και στην προηγούμενη θητεία με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνει ένα ψήφισμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απορώ που το γραφείο ευρεσιτεχνιών δεν κάνει αυτό που το ίδιο θεωρεί ότι είναι το σωστό και φαίνεται να ακολουθεί άλλες πολιτικές κατευθύνσεις. Ε, ίσως ε, ο λόγος μπορεί να αναζητηθεί στο γεγονός ότι το γραφείο αυτό ζει από την χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Γι' αυτό και ενδεχομένω έχουν μια δική τους δυναμική. Ε, έχουν ε, λόγο βεβαίως να θέλουν για όλα, για όλα τα πράγματα που θα μπορούσαν να εκδοθούν ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας να εκδίδονται τέτοια. Εμείς όμως έχουμε τελείως διαφορετικό ρόλο. Θα ήταν πολιτικό σκάνδαλο να εγκρίνουμε κάτι τέτοιο για βιολογικές διεργασίες να δίνονται δηλαδή πατέντες. Ε, δεν ξέρω ποιο ακριβώς βρίσκεται πίσω ε, από την όλη ιστορία. Ε, είναι πραγματικά περίεργο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κομισιόν να συμφωνούν και να μην μπορούν να επιβάλλουν στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, την δική τους θέση. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς μα κοροϊδεύει. Ε, έρχεται τώρα για τρίτη φορά το καθήκον να εγκρίνουμε άλλο ένα ψήφισμα, τι θα γίνει, θα έχουμε και κάποιο τέταρτο στο άμεσο μέλλον ας πούμε. Νομίζω ότι κάποιο επιτέλους πρέπει να επιβληθεί, να επιβάλλει τη θέση του στο γραφείο Εύρεσης Τεχνιών, ε, γιατί δεν μπορεί αυτό το γραφείο ε, να ενεργεί ενάντια σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πολιτικές κατευθύνσεις που έχουν δοθεί. Νομίζω ότι αυτό ε, είναι απαράδεκτο Μπορούμε βεβαίω ε, να εγκρίνουμε το ψήφισμα, να κάνουμε και μια γνωμοδότηση, αλλά νομίζω ότι είναι σαφέ ότι δεν μπορεί να σηκώνει ε, μπαϊράκι έτσι μόνο του και αυτόνομα το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία. Ευχαριστώ, ο κύριο Φλάναγκαν. Um, uh, ναι, Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα βρει κανείς Ευρωπαίο ψηφοφόρο που θα συμφωνήσει με την ιδέα ότι μπορούν να πατενταριστούν βιολογικές διαδικασίες. Γι' αυτό και προφανώς και πρέπει να εγκρίνουμε αυτό το ψήφισμα. Αυτό που είπε ε, και ο συνάδελφος Χόισμαν είναι ότι αυτές, ε, αυτές οι υποθέσεις δεν θα πρέπει να βρίσκονται στα χέρια λίγων. Συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη θέση και ε, οι διαδικασίες ε, ε, γενετικής τροποποίησης βιολογικών έχουμε εμπειρία πλέον ότι τελικά ωφελούν τους λίγους και όχι τους πολλούς. Εμείς είμαστε ιδιοκτήτες όλης αυτής της γνώσης. Ακόμη και οι πατέντες που έχουν δοθεί ε, βασίζονται σε γνώση που έχει αποκτηθεί μέσα από τα εκπαιδευτικά συστήματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από τους φορολογούμενους δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κάποιου να θεωρούν ότι αυτή η γνώση του ανήκει και μάλιστα να κερδοφορούν ε, ει βάρο ε, των πολλών. Ε, δεν είναι δυνατόν να είναι ατομική ιδιοκτησία ορισμένων λίγων οι βιολογικέ διεργασίε. Ευχαριστώ πολύ ο συνάδελφος Ρούσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον συνάδελφο Χόιτεμα που έθεσε αυτό το σημαντικό θέμα. Και εγώ συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Είναι πολύ σημαντικό ως Επιτροπή Γεωργίας να αποφανθούμε σαφώς επί αυτού και προσυπογράφω και εγώ. Ήρθε πια η ώρα να κλείσουμε αυτό το νομοθετικό παραθυράκι. Έχω την εντύπωση ότι όλοι συμφωνούμε για την ανάγκη αυτή. Όλοι συμφωνούμε ότι το φυτικό υλικό ε, μέσα από κυρίως βιολογικές μεθόδους δεν πρέπει να κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η οδηγία άλλωστε δεν είχε αυτό το νόημα. Το φυτικό υλικό πρέπει να παραμένει ελεύθερα προσβάσιμο στους βελτιωτές φυτών για να μπορούν να αναπτύσσουν νέες ε, καλές ποικιλίε. Και το Κοινοβούλιο ε, ήταν απόλυτα ξεκάθαρο κατά την προηγούμενη θητεία του και η θέση της Κομισιόν ήταν ξεκάθαρη επίσης. Τα μέλη του Γραφείου Βρεσιτεχνιών είπαν ότι θέλουν να κλείσουν αυτό το κενό. Το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να προχωρήσουμε στα διοικητικά βήματα και να ε, καταρρύψουμε αυτό το εμπόδιο στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών. Αν γίνει αυτό θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα για να κάνουμε αυτή τη βασική δήλωση ότι το φυτικό υλικό δεν πρέπει να κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ευχαριστώ και πάλι τον συνάδελφο Χόιτεμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μπούντα, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τον συνάδελφο για την πρωτοβουλία. Δεν θα πρέπει εμείς ε, να είμαστε οι κάθε φορά που γίνεται περκαγιά. Και φυσικά οι διαδικασίες δεν μπορεί να είναι αντικείμενο διπλώματος ευρεσιτεχνία. Αυτό είναι αυτονόητο. Και οι συνέπειες ήταν καταστροφικές αν επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Όχι μόνο για τους Γιώργους, που θα πρέπει να καταβάλουν πολύ περισσότερα χρήματα για να χρησιμοποιήσουν τέτοιες ε, πατενταρισμένες ποικιλίε, αλλά σκεφτείτε πόσο δένουμε τα χέρια και των ερευνητών. Και έχουμε και το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών. Αλλά ας μην ξεχνάμε και τους καταναλωτές. Και αυτοί θα χρειαστεί ε, να πληρώσουν μεγαλύτερο τίμημα για τέτοια προϊόντα που καλύπτονται από πατέντες. Κύριε Μακιντάιρ. Ευχαριστώ. Κι εγώ συμφωνώ και υποστηρίζω και είμαι και ευγνώμων στον Γιάννο Χοίτεμα που έθεσε το θέμα αυτό. Δύο πράγματα θα πω. Συμφωνώ με όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι σήμερα, αλλά αν με δίπλωμα ευρεσιτεχνία, τι πρέπει να κάνουμε. Θα δείξουμε μια εφεύρεση, ένα βήμα εφεύρεσης. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν πρόκειται για μια κυρίως βιολογική μέθοδο. Πώς μπορεί να είναι θέμα που να, συνε... να, σημαίνει και εφεύρεση. Δεν μπορεί λοιπόν να ε, καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το ζωικό και φυτικό υλικό να παραμένει ανοιχτό στους βελτιωτές ε, φυτών και ζώων για να επιλέγουν ε, στις ε, πιο ανθεκτικές ποικιλίε. Και μιλήσαμε πολύ στο παρελθόν για την ανάγκη ε, γενετικής ποικιλότητα και την ανάγκη ύπαρξης μεγάλου γενετικού υλικού και μιας δεξαμενής γενετικής ε, ανοιχτά προσβάσιμη σε όλους. Θα με ανησυχούσε πάρα πολύ αν οι μικροί βελτιωτές και οι μικροί γεωργοί ξαφνικά έβλεπαν ότι το γενετικό αυτό υλικό δεν τους είναι προσβάσιμο γιατί κάποιος ε, αξίωσε ευρεσιτεχνία. Ε, νομίζω ότι υπάρχει διαπαραταξιακή συμφωνία εδώ και μου που Ευχαριστώ. Κρίστενσεν. Χωρίς μικρόφωνο. Θα μιλήσω στα δανέζικα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάνν Χόιτεμα για την πρωτοβουλία του. Ευχαριστώ που άρχισατε αυτή τη συζήτηση. Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του συναδέλφου. Μιλάμε για μεγάλα οικονομικά συμφέροντα εδώ, πολυεθνικές ε, εταιρείε που θέλουν να, να κατοχυρώσουν ευρεσιτεχνίες. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Και μην ξεχνάμε και το θέμα της δημόσιας υγείας και τα ευρύτερα θέματα υγείας που λέγουν όχι στην ε, κάλυψη με ευρεσιτεχνία αυτών των ε, ζώντων οργανισμών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Ευχαριστώ. Η εμπειρία μου ε, είναι από τα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία ε, καλύπτονται από ευρεσιτεχνίες και υπάρχουν κάποιες παραλληλίες εδώ. Πρώτον, δεν πρέπει να επιτρέπεται να Υπάρχουν ποικιλίε με βρεσιτεχνίες ε, όταν ήδη αυτές υφίστανται. Αυτό είναι προφανές, είναι αυτονόητο. Από την άλλη πλευρά, ακόμα και αν λέμε ότι αυτές οι ποικιλίε προέρχονται από κυρίως βιολογικές μεθόδους, ε, όμως η βελτίωση έχει κάποιο κόστος και αν θέλει κάποιος να επενδύσει στη βελτίωση νέων φυτικών ποικιλιών θα πρέπει να υπάρχει κάποια διασφάλιση ότι για κάποιο χρονικό διάστημα και το ίδιο ισχύει και για τα φαρμακευτικά προϊόντα θα πρέπει να θα μπορεί κανείς Βέβαια μπορεί κανείς να παρατείνει επάπειρον την ε, ε, περίοδο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια περίοδος περιορισμένη όπου θα υπάρχουν αποκλειστικά δικαιώματα και θα ε, υπάρχει απόδοση των επενδύσεων που έγιναν και υπάρχουν ε, βελτιωτές που θα, θα, έχουν ένα πλεονέκτημα και θα μπορεί να ενθαρρυνθεί έτσι η ε, βελτίωση των ποικιλιών. Αν λέμε δηλαδή ε, έτσι ε, γενικά ότι δεν μπορούμε να δώσουμε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αυτό είναι λάθος. Γιατί αν δεν, ε, καλό θα ήταν να μπορούμε να διασφαλίσουμε τη, τη, τη νέα αυτή ποικιλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μπίτο. Και ευχαριστώ τον κύριο Χαϊτομα για την πρωτοβουλία του. Και αυτή η ιδέα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας φυτών που είναι αποτέλεσμα βιολογικής διεργασίας ε, ουσιαστικά θέλει να κατάσχει το, τη γενετική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Μιλούμε για ε, πανάρχες διαδικασίες. Ο πρώτος ε, βελτιωτής ε, φυτών, δημιουργός ε, ποικιλία είναι ο Γιώργος. Ήταν, είναι και θα είναι ο Γιώργος. Είναι τεράστιες, ε, τεράστια τα δικηβεύματα αυτής της υπόθεσης και μάλιστα συνδέονται με κάτι άλλο που είναι της επικαιρότητα, η αυτονομία του αγρότη για, τους ε, γενετικούς για, τους για το γενετικό υλικό, για τους σπόρους και αν θα πρέπει ο Γεωργός να χρησιμοποιεί μόνο τους σπόρους που ο ίδιος ε, συνέλεξε, φανταστείτε την καταγραφή που θα δημιουργηθεί. Να τον υποχρεώσουμε να χρησιμοποιεί μόνο σπόρους που ο ίδιος καλλιέργησε και ο ίδιος ε, ε, παρήγαγε, αποκλείεται. Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση στις κλιματικές αλλαγές είναι η προσαρμογή των γενετικών πόρων με τους οικοτύπους, όπως λέμε, δεν θέλω να επισέλθω σε τεχνικά θέματα, ώστε να έχουμε μια εξέλιξη του γενετικού πόρου ανάλογα με την εξέλιξη του ε, περιβάλλοντος, κλιματική ή άλλη εξέλιξη. Οπότε προσχωρώ και εγώ σε αυτή τη λογική και ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Χαίτημα που επανέφερε αυτό το θέμα στην ε, ημερήσια διάταξη γιατί αν επιτρέψουμε κάτι τέτοιο ουσιαστικά θα αντισταθούμε στο ορού της ιστορίας και είναι τεράστια τα δικηβεύματα και για τις ε, σημερινές αλλά και για τις επερχόμενες γενιές. Ωραία. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει συνένεση. Θα δώσω όμως το λόγο στην Κομισιόν για να μας μιλήσει για τα διαδικαστικά. Ποιες είναι οι δικές μας αρμοδιότητες, ή για να μας ε, δώσει τη δική της εκτίμηση για το τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή, Επιτροπή Γεωργίας, πώς θα πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα και ως Επιτροπή και ως ε, μεμονωμένοι Ευρωβουλευτές. Ας μας τα πει όλα αυτά η Κομισιόν. Παρακαλώ. Um, yes, hi. Um, thank um, Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Με βάση τους κανόνες της συνθήκης και μιλώ με την ιδιότητα της ε, αξιωματούχου της υπηρεσίας μου, η Κομισιόν βεβαίως εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διευρωμένο Συμβούλιο. Αν θέλουν όμως και ε, μεμονωμένα άτομα να υποβάλουν σχόλια. Αυτό έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Και αυτό βεβαίω ισχύει και για ευρωβουλευτέ. Όπω γνωρίζετε, εμεί ω Κομισιόν έχουμε συντάξει ένα σημείωμα. Η Κομισιόν επίσης πρόσφατα ε, το υποστήριξε το σημείωμα και βλέπετε ότι ε, έχουμε υποστηρίξει και ενώπιον του διευρυμένου συμβουλίου ε, το σημείωμα αυτό. Οπότε είναι προφανές ότι εμείς ε, από την πλευρά μας θα υποστηρίξουμε κάθε άλλον ε, φορέα ή μεμονωμένο άτομο που θα τοποθετηθεί με παρόμοιο τρόπο με τον οποίο τοποθετούμαστε και εμείς. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Χόιτεμα, θέλετε το λόγο. Δεν ξέρω αν, συμφωνείτε δηλαδή και, σε, και πέραν της Επιτροπής να αναλυθούν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Να, να το ξεκαθαρίσω λίγο. Εμείς ως μεμονωμένα μέλη τη Επιτροπή, εντάξει, το είπε και η Κομισιόν ότι μπορούμε ενδεχομένως να τροφοδοτήσουμε την γενικότερη συζήτηση που θα γίνει στο Γραφείο ε, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία. Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά για να ασκήσουμε ακόμη μεγαλύτερη πίεση μπορούμε να εγκρίνουμε και εμεί ένα ψήφισμα. Δεν θα τροφοδοτήσει ακριβώς τη συζήτηση στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών, όμως θα είναι μια πολιτική τοποθέτηση ε, που θα λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμφωνεί ε, με μια τέτοια πρακτική που πάει να κατοχυρωθεί στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών. Κύριε Τσόλος, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν αρκούν ε, οι προσωπικές απόψεις κάποιων ευρωβουλευτών. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο, ένα κατηγορηματικό και ξεκάθαρο μήνυμα του Νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπε και ο συνάδελφος Μπούντα, θα πρέπει να στείλουμε ένα περίφραστο μήνυμα ε, διατρανώνοντα την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Δεν είναι μόνο νομικό το ζήτημα, είναι και ηθικό, δεοντολογικό θέμα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύσσωμο και όχι μόνο από νομομαθήσει από δικηγόρους στη συζήτηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να στείλουμε ένα περίφραστο μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του θεσμικού οργάνου που είναι άμεσα εκλεγμένο από του Ευρωπαίου πολίτε και να μην έχουμε μόνο το μήνυμα ενό θεσμικού οργάνου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να το εξηγήσω λίγο. Ε, επί της ουσίας συμφωνούμε. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ένα ψήφισμα θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς δεν μπορούμε πριν από την προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου να καταλήξουμε στην έγκριση ενός τέτοιου ψηφίσματος. Την μεθεπόμενη εβδομάδα έχουμε ολομέλεια που θα ήταν η μοναδική ευκαιρία να υποβληθεί και να εγκριθεί ένα τέτοιο ψήφισμα. Και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει μέσω της Επιτροπής ε, Γεωργίας, θα μπορούσε όμως μέσω των πολιτικών ομάδων, έτσι μου λέει η γραμματεία της Επιτροπής μας. Δηλαδή όχι από τη δική μας Επιτροπή να ξεκινήσει αυτό το ψήφισμα, αλλά από τις πολιτικές ομάδες και να ε, υποβληθεί στην Ολομέλεια ένα τέτοιο σχέδιο ψηφίσματος. Αυτή είναι η δυνατότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ε, όχι όμως από την Επιτροπή Γεωργίας ώστε να προλάβουμε και την προθεσμία τη 1 η Οκτωβρίου. Ο κύριο Χόισλερ. Ε, εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να τοποθετηθούμε μονομένα ως Ευρωβουλευτές, αλλά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, δεν νομίζω ε, ότι οι πολιτικές ομάδες ε, ε, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Μπορούν να το κάνουν, να υπάρξει και ένα τρίτο ψήφισμα και εναπόκειται μετά στην ε, διάσκεψη των Προέδρων για να υποβληθεί στην Ολομέλεια ένα τέτοιο ψήφισμα για να στείλουμε και ένα σαφές μήνυμα. Ε, δεν νομίζω ότι ε, θα είχε και νόημα ε, εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας απλώς να στείλουμε ε, ένα μήνυμα. Χρειαζόμαστε όλο το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι σε αυτό, αφού συμφωνούν και όλες οι πολιτικές ομάδες, είναι κάτι το εφικτό, μπορεί να γίνει, οπότε μπορούμε να προσπαθήσουμε μέσω των πολιτικών ομάδων να πιέσουμε ώστε να μπει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η προσπάθειά μας. Ευχαριστώ. Κυρία Μιλό, συμφωνώ με τον συνάδελφο. Αν συμφωνούν όλες οι ομάδες και συζητηθεί το θέμα σε όλες τις ομάδες, η πρόταση ψηφίσματος μπορεί να συνταχθεί χωρίς κανένα πρόβλημα και διαπαραταξιακά να συζητηθεί το θέμα στην επόμενη Ολομέλεια. Θα είναι ξεκάθαρο το μήνυμα και θα είμαστε και μέσα στα χρονικά περιθώρια. Εντάξει. Ο συνάδελφος Σιόλος πάλι. Εγώ είμαι έτοιμος να το προτείνω αυτό στη διάσκεψη των Προέδρων. Αν ε, με στηρίζουν όλες οι ομάδες, θα συνεννοηθώ με τους επικεφαλείς των ομάδων και θα το συζητήσουμε στη διάσκεψη των Προέδρων για να ληφθούν μέτρα από το Κοινοβούλιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να δρούμε προορατικά. Ευχαριστώ, ο συνάδελφος Δεκάστρο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ακολουθώντας το συλλογισμό του Dutch Solos θα έστελνα σε όλες τις ομάδες της Επιτροπής, ε, από όλες τις ομάδες της Επιτροπής, ε, επιστολή προς τη διάσκεψη των Πρόεδρων ζητώντας να μπει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πιο ισχυρό μας ε, μέσο για άσκηση επιρροής. Okay, Καλώς. Η Κομισιόν ζήτησε και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ. Μια σύντομη διευκρίνηση. Πολιτικό ψήφισμα είναι επιλογή του Κοινοβουλίου προφανώς και θα είναι και πολύ καλή υποστήριξη για την υπόθεση. Για το χρονοδιάγραμμα όμως, γιατί είπατε το 1η Οκτωβρίου προθεσμία, αν είναι μετά το ψήφισμα πρέπει να ξέρετε ότι συνήθως οι διαδικασίες μπροστά στο Διευρυμένο Συμβούλιο Προσφυγών ε, παίρνουν 20 μήνες περίπου για να γίνει διαδικασία. Δεν νομίζω ότι θα καθυστερήσετε λοιπόν ακόμα και αν, ή, το, το ψήφισμα γίνει δεκτό μετά την προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου. Η 1η Οκτωβρίου είναι μια διαδικαστική προθεσμία για να γίνει προσφυγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πολιτικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου είναι χρήσιμο είτε ε, είναι της 1 η Οκτωβρίου ή 10 μέρες μετά ή και 10 μήνες μετά. Δεν ε, θα κρίνει το Συμβούλιο, ε, σίγουρα όχι δεν θα κρίνει φέτος. jetzt Καλά. Έχουμε τώρα διαφορετικές προτάσεις. Ε, ήταν λίγο διαφορετική η πρώτη δήλωση της Κομισιόν, οπότε καλή είναι η διευκρίνηση που δόθηκε τώρα, ότι δηλαδή το ψήφισμα μπορεί να ισχύει και μετά. Δύο εναλλακτικές λοιπόν, είτε τη διαδικασία μέσω της, της Επιτροπής μας ή η ταχύτερη διαδικασία για την επόμενη Ολομέλεια. Το ερώτημα είναι, θα αποφασίσουμε τώρα ή θα συζητηθεί και πάλι από τους συντονιστές για να συμφωνήσουμε επί της διαδικασίας. Η κυρία Μούλερ, ε, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, για το κοινοβούλιο, για, για, για, τα ευρωπαϊκά όργανα, ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό το κοινοβούλιο ως ερετό που έλαβε θέση διαπαραταξιακά να ε, δράσει αντιμετωπίζοντας το θέμα ως κατεπήγον. Πριν από την 1η Οκτωβρίου λοιπόν θα έπρεπε να περάσει το ψήφισμα. Είναι ξεκάθαρα τα ζητήματα, ξέρουμε που, τις θέσεις όλων. Γιατί λοιπόν να επιλέξουμε μια μακρόχρονη διαδικασία ενώ μπορούμε να διαλέξουμε μια συνοπτική. Ο κύριος Στόρφαν, η συζήτηση εδώ έδειξε ότι συμφωνούμε όλοι. Προτείνω αυτό και εγώ αυτό που είπες να συζητηθεί και από τους συντονιστές ε, τι είναι το καλύτερο να γίνει από το Κοινοβούλιο, τι ανταποκρίνεται καλύτερα στα δικά μας τα συμφέροντα και να συνεχίσουμε. Κύριο κύριος Αντριέ. Ναι, αλλά θα πρέπει να σπεύσουμε, γιατί υπάρχει ομοφωνία, φαίνονται απλά τα πράγματα. Και νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη πρόταση του κυρίου Παύλου Τικάστρο να στείλουμε επίσημη επιστολή στη διάσκεψη των Προέδρων, ζητώντα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει θέση σε επίπεδο ολομέλεια. Θα πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Γιατί, όπω είπε και ο Ντάτσαν η, θέση μα είναι ξεκάθαρη και το διακύβευμα είναι και διοντολογικό ηθική φύση. Κυρία Πίρικ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την τελευταία παρατήρηση. Κυρία Μίλλερ, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να προωθήσουμε το θέμα, γιατί περιμέναμε ήδη πολύ καιρό. Θέλουμε απόλυτη σαφήνεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφής, αλλά υπάρχουν κάποιοι και οργανώσεις που έχουν αντίθετα συμφέροντα οι απόψει. Εμείς θα πρέπει να διατρανώσουμε το δικό μας μήνυμα. Ο συνάδελφος Χόιτμαν θέλει το λόγο. Ναι, εγώ είμαι λίγο πιο ρεαλιστής. Για μένα η προθεσμία της 1ης ε, Οκτωβρίου δεν είναι τόσο ιερή. Πιο σημαντικό είναι να, έχουμε, να εμφανιστούμε πραγματικά με μια φωνή και να ασκήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά. Αλλά ας το αποφασίσουν και οι συντονιστές βεβαίως. Λοιπόν, συμφωνείτε να συζητηθεί το θέμα στους συντονιστές αμέσως μετά την ε, συνεδρίασή μας στη βάση της ε, πολιτικής βούλησης που εκφράστηκε που είναι ενιαία και ομόφωνη. Είναι δευτερεύοντο ζήτημα το διαδικαστικό του πώς θα προχωρήσουμε δηλαδή. Ωραία, αφού δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα διακόψουμε τη συνεδρίασή μας. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διάταξης για την πρωινή συνεδρίαση μιλώ. Τώρα το, μόνο ερώτημα που απομένει είναι θέλετε να ξεκινήσουμε αμέσως με τη συνεδρίαση των συντενιστών ή θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 11. Εγώ ε, είμαι ανοιχτός Τώρα. Να την κάνουμε τώρα. Ωραία. Πέντε λεπτά διαλυματάκι και συνεχίζουμε αμέσως μετά με τη συνεδρίαση των συντονιστών.